Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας καλωσορίσω στη συνεδρία της Επιτροπής μας σήμερα. Να καλωσορίσω επίσης όλους τους εκπροσώπους των διπλωματικών αποστολών, την αυτού εξοχότητα των πρέσβη της Νικαράγουα, κύριο Σαντίνο, την αυτού εξοχότητα πρέσβη του Ελ την κυρία Βιλατότο, θα ήθελα επίση να καλωσορίσω όλους τους εκπροσώπους τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Πόνς, αναπληρωτή προϊστάμενο διεύθυνση για την Κεντρική Αμερική, το Μεξικό και την Καραϊβική της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, τον κύριο Κοστέλο, προϊστάμενο της Διεύθυνσης των Εκλογικών Παρατηρητών της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Η διερμηνία θα παρέχεται στην Αγγλική, Ισπανική, Ελληνική και Παθητική στα Γαλλικά. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το διαδίκτυο το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης σας έχει διανεμηθεί στα αγγλικά, στα ελληνικά και στα ισπανικά και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα θεωρηθεί ότι η ημερήσια διάταξη έχει εγκριθεί. Τα πρακτικά της συνεδρίας της 4 Φεβρουαρίου του 2017 περιλαμβάνονται στο φάκελο που σας έχει διανεμηθεί και αν δεν υποβληθούν τροποποίησεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα εγκριθούν χωρίς αλλαγή ή εάν γίνουν κάποιες αλλαγές θα συμπεριληφθούν και αυτές. Να πάμε τώρα στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, που είναι, έχει να κάνει με την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογών της 26 Νοεμβρίου 2017 στην Ονδούρα. Κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, η Ονδούρα πραγματοποίησε γενικές εκλογές τον Νοέμβρη του περασμένου χρόνου, οι πολίτες της Ονδούρα κλήθηκαν να εκλέξουν νέο πρόεδρο, 128 νέα μέλη για το Εθνικό Κογκρέσο, 20 μέλη για το Κοινοβούλιο της Κεντρικής Αμερικής, καθώς και νέους δημάρχους για τους Δήμους της Ονδούρας. Η προεδρική εκλογή ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε μετά την τροποποίηση του συντάγματος της Ονδούρας, επιτρέποντας τον ενεργεία πρόεδρο να επιδιώξει την επανεκλογή του. Όπως γνωρίζετε, η απόφαση αυτή δημιούργησε έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, καθώς η δυνατότητα αλλαγής του συντάγματος με σκοπό την προεδρική επανεκλογή ήταν η πρωταρχική αιτιολογία για την απομάκρυση του Προέδρου Ζελάγια από το αξίωμα το 2009. Τα αρχικά αποτελέσματα της εκλογικής ψηφοφορίας έδιναν ένα σημαντικό προβάδισμα στον υποψήφιο της αντιπολίτευσης κ. Νασράλα, Στη συνέχεια η δημόσια ενημέρωση για την καταμέτρηση διακόπτηκε για περισσότερο από μία ημέρα και με την αποκατάσταση της ροής πληροφόρησης η διαφαινόμενη επικράτηση του υποψηφίου Προέδρου Νασράλα άρχισε να μειώνεται σταδιακά και τελικά ο πρόεδρος Χερνάντες επικράτησε στις καταμετρήσεις εκλογικής ψηφοφορίας εν μέσω πολυάριθμων καταγγελιών για παρατυπίες που οδήγησαν σε έντονες διαμαρτυρίες για εκλογική νοθεία και σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα κατά την διάρκεια των οποίων τουλάχιστον 17 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Με την ολοκλήρωση εκλογικής διαδικασίας και οι δύο υποψήφοι ισχυρίστηκαν ότι νίκησαν. Στις 17 Δεκεμβρίου, 21 μέρες μετά την εκλογική αναμέτρηση, το ανώτατο εκλογικό δικαστήριο ανακήρυξε νικητή τον πρόεδρο Χερνάντες με ποσοστό 42,95% επί του συνόλου των ψήφων έναντι 41,4% του υποψηφίου Νασράλα. Ωστόσο, η αποστολή εκλογικής παρατήρησης του Οργανισμού Αμερικανικών Χωρών σημείωσε στην προκαταρκτική της έκθεση ότι η εκλογική διαδικασία χαρακτηρίστηκε από παρατυπίες και ελλείψεις, χαμηλή τεχνική ποιότητα και απουσία κυριότητας και ζήτησε να πραγματοποιηθούν νέες εκλογές. Η αντιπροσωπεία μας περιμένει με ενδιαφέρον να δει και τα τελικά συμπεράσματα των αποστολών εκλογικής παρατήρησης του Οργανισμού Αμερικανικών Χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι ιδιαίτερα που η επικεφαλής της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Ματίας, αποδέχθηκε την πρόσκληση της αντιπροσωπείας μας για να ενημερώσει τα μέλη της ΔΕΚΑΜ σχετικά με τα συμπεράσματα της αποστολής. Θα ήθελα λοιπόν, κυρία Ματίας, να σας δώσω το λόγο για την ενημέρωσή μας. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη σε αυτά που θα πω, παρόλο που η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη. Αν ε, μιλήσω περισσότερη ώρα από όσο έχεις προβλέψει, κάνε μου ένα νεύμα για να συντομεύσω. Μιλάω εκ μέρους Τη αποστολή Παρατηρητών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν έχουμε ακόμα την τελική μα έκθεση, αλλά θα προσπαθήσω να οργανώσω τι σκέψει μου γύρω από τρει άξονε Πριν τι εκλογέ πρώτον, η μέρα των εκλογών και μετά τι εκλογέ. Όπω είπε και εσύ στην εισαγωγή σου, όντω ήταν πολύ επίμαχο το θέμα τη εκλογική διαδικασία. ήδη και υπήρξαν πράγματα τα οποία δεν βλέπονταν από το Σύνταγμα, αλλά που ευετράπησαν στη συνέχεια. Ήταν περίπλοκη η κατάσταση και η διαδικασία, πράγματα τα οποία συζητήθηκαν πάρα πολύ και εκτός από αυτά πρέπει να πω ότι όταν αποφάσισαν όλοι τα κόμματα να συμμετάσχουν στις ε, εκλογές, αυτό επικυρώθηκε από τους διάφορους ε, φορείς, εγκρίθηκε και η δικιά μας αποστολή παρατηρητών, γι' αυτό και πήγανε. Είχαμε μια πρώτη προκαταρτική έκθεση που βασίζεται στα στοιχεία που έχουμε από την περίοδο πριν των εκλογών. Ξέρετε ότι κράτησε πολύ η παρατήρηση, αλλά υπήρχε και ένα πιο σύντομο διάστημα το τελευταίο καιρό. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, είναι πράγματα γνωστά, θα περάσω στο περιεχόμενο. Στη διαδικασία αυτή της μακράς διάρκειας παρατήρηση αλλά και της προκαταρτικής έκθεσης που έχουμε ετοιμάσει εντοπίσαμε διάφορα πράγματα. Κάποια από αυτά είχαν παρατηρηθεί και το 2013 στις εκλογές και κάποια άλλα είναι νέα. Η επανεκλογή πρώτα απ' όλα που ήταν το επίμαχο ζήτημα, το κυρίως επίμαχο ζήτημα. Μπορέσαμε Πάντως ε, να πούμε ότι δεν υπήρξε και πλήρης ανεξαρτησία όσον αφορά τα εκλογικά δικαστήρια, αλλά και του συνταγματικού σώματος. Μιλήσαμε επίσης και για επιρροές εγκληματικών οργανώσεων ουσιαστικά που δρούν και σε άλλες χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Αναφέραμε επίσης όσον αφορά την προεκλογική εκστρατεία, όσον αφορά το χώρο που δόθηκε, η δυνατότητα ε, παρεμβάσεων ε, στη τηλεόραση κλπ. Διαπιστώσαμε ότι ο τωρινός πρόεδρος είχε 86% του διατηθέμενου χρόνου, ενώ μόνο 6% υποψήφιο τη αντιπολίτευση. Και μιλάμε για τη δημόσια τηλεόραση εδώ, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα τα αναφέραμε, δώσαμε τα στοιχεία στα παραρτήματα και βλέπετε στην προκαταρτική μας ε, έκθεση ότι όλα αυτά έχουν δημοσιευτεί. Επίσης, οι πόροι δεν ήταν σε καλή ισορροπία, δηλαδή πόσα χρήματα πήρε ο κάθε υποψήφιος για την προεκλογική του εκστρατεία και βέβαια το Εθνικό Κόμμα, το κόμμα του τέος και τωρινού Προέδρου ήταν αυτό που βγήκε κερδισμένο. Όσον αφορά την εκλογική διαδικασία την ημέρα των εκλογών. Αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ότι καλά οργανωμένες οι εκλογές δεν υπήρξαν ιδιαίτερα επεισόδια, συμβάντα. Φαινόταν να διεξάγονται όλα κανονικά. Δεν εντοπίστηκαν ιδιαίτερα θέματα βίας ή αδυναμία των ανθρώπων να πάνε να ψηφίσουν εκτός από τις περιοχές εκείνες όπου κυριαρχούν οι Μάρας. Αυτό που διαπιστώσαμε επίσης ήταν κάποια μικρά προβληματάκια, τίποτα όμως που να υπονομεύει πραγματικά την εκλογική διαδικασία αυτή καθεαυτή. Μετά όμως άρχισαν τα επίμαχα ζητήματα ότι υπήρξε υπόσχεση ότι τα αποτελέσματα ε, θα δημοσιευθούν αμέσως, θα δοθούν ε, στη δημοσιότητα. Αυτό όμως δεν έγινε, παρόλο που το είχαν υποσχεθεί. Δημιουργήθηκε σύγχυση Και όχι μόνο αυτό, αλλά και δυσπιστία. Γιατί για πολλές ώρες δεν υπήρξε απευθεία ε, αναμετάδοση. Και όταν ε, υπήρξε και πάλι σύνδεση, διαπιστώσαμε ότι είχε αλλάξει το αποτέλεσμα, ότι δηλαδή η δύναμη του Ναστράλα, του υποψήφιου της ε, αντιπολίτευσης μειωνόταν και η διαφορά μεγάλωνε. Και κάθε φορά μετά από τη διακοπή διαπιστώναμε νέα εξέλιξη και διαφορά πάλι στα αποτελέσματα. Και έτσι τελικά ο προηγούμενος ε, πρόεδρος και ο τωρινός ε, όταν ε, ξανά μπαινε προς το σύστημα φαινόταν να κερδίζει. Στη συνέχεια έλαβε χώρα πολλές διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες. Εμείς καταδικάσαμε φυσικά τη βία, την καταπίεση που έλαβε χώρα αυτές τις επόμενες μέρες, ακόμα και το κράτος έκτακτης ανάγκης το οποίο προκήρυξε ο πρόεδρος τότε. Διαπιστώσαμε ότι υπήρξαν πολλές προσφυγές όσον αφορά τις δημοτικές και τις κοινοβουλευτικές εκλογές, ενώ εμείς ήμασταν παρατηρητές εκεί κυρίως για τις προεδρικές. Οι προσφυγές που έγιναν στο Νότο Εκλογικό Δικαστήριο δεν υποβάλλονταν με αρκετές αποδείξεις. Οπότε χρειάστηκε χρόνος για να διαπιστώσουμε τι έχει γίνει με την καταμέτρηση. 5.000 ψηφοδέλτια δεν πήγανε από τα εκλογικά κέντρα Άρα χρειάστηκε να ξαναγίνει καταμέτρηση και για αυτά για τα οποία γίνονταν οι προσφυγές. Υπήρχαν βέβαια και αυτό που σας είπα που χάθηκαν, δεν μπορέσαμε να τα μετρήσουμε. Πάντως αυτό που μπορώ βασικά να πω είναι ότι 80% πήραμε από τα διάφορα εκλογικά τμήματα, τα πεπραγμένα τους τουλάχιστον, αλλά όχι όλα. Και τα πήγαμε στο σταγματικό δικαστήριο. Ήταν εντελώς διαφορετικά τα αποτελέσματα τα οποία φτάσαν από τα εκλογικά κέντρα και τα αποτελέσματα τα οποία τελικά διαπιστώναμε ότι είχαν ανακοινωθεί. Εμείς και το ξέρουν και μέλη του Κοινοβουλίου, ήμασταν παρατηρητές θέλοντας τη διαφάνεια, αλλά διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν διαφορές στις πηγές που είχαμε στη διάθεσή μας και ότι υπήρχαν και προβλήματα στην προεκλογική εκστρατεία. Πάντως για τα αποτελέσματα αυτά, καθεαυτά αυτά, για την καταμέτρηση, τελικά μεταξύ μας δεν βρήκαμε διαφορές και τα τρία κύρια κόμματα μας δώσανε όλα τα προηγούμενα. αλλά όπως σας είπα μόνο το 80% μας δώσανε. Δεν μπορέσαμε να έχουμε πραγματικά αντίγραφα χωρίς αποδείξεις. Δεν μας διευκολύνουν τη ζωή βέβαια γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν γίνονται προσφυγές για κάποια στοιχεία και εμείς δεν έχουμε αποδείξεις για το τι δεν πήγε καλά ή ότι πήγε καλά, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Και τα ξέρουμε αυτά και από την προηγούμενη αποστολή παρατηρητών. Λοιπόν, τώρα, τι γίνεται. Καμία από τις προσφυγές δεν οδήγησε σε επανακαταμέτρηση. Γιατί καμία προσφυγή δεν ζητούσε ούτε μερική ούτε πλήρη νέα καταμέτρηση. Μόνο προσφυγές υπήρχαν που ζητούσαν ε, να ε, κρυθεί άκυρη η εκλογή του Προέδρου, χωρίς όμως αποδείξεις πάλι. Ε, η στιγμή είναι δύσκολη, ανέλαβε ο πρόεδρος. Εξακολουθούν να γίνονται πολλές ε, διαδηλώσεις, να υπάρχουν υψηλά επίπεδα βίας και καταστολής, που εννοείται ότι καταδικάζουμε και το έχουμε ήδη κάνει. Θα έχουμε σύντομα την τελική μας έκθεση και θα επιστρέψουμε στη χώρα, στην Οδούρα, για να παρουσιάσουμε την έκθεσή μας αυτή με εντολή διαφορετική από εκείνη της ε, υπηρεσία εξωτερική δράσης που είναι μια ανάμειξη και πλήρη σεβασμού του διεθνού δικαίου. Βάσει αυτών θα είναι η τελική μας έκθεση και ευχαρίστω να ξαναέρθω να σας πω περισσότερα τότε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, ενημέρωση. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι γι' αυτό εξοχότητα ο πρέσβης της ονδούρα ο κύριος ε, Οτσόα, δεν μπορεί να παραστεί σήμερα και ζήτησε να κάνει μια μικρή δήλωση ο κύριος Ατάλα από την ε, Πρεσβεία. Κύριε Ατάλα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε εκ μέρου ε, τη ε, αντιπροσωπεία ε, τη Ονδρό στην Ένωση. Σα ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην χώρα μα και η αποστολή εκλογική παρατήρηση. Πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρουσία τη εκεί υπό την χεισέ τη κυρία Ματία. Ήταν μια αντιπροσωπεία που έδειξε επαγγελματισμό, αμεροληψία, αντικειμενικότητα. Γνωρίζουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλέ προκλήσει και γνωρίζουμε νομίζουμε ότι τώρα θα πρέπει να υπάρξει η εθνική συμφιλίωση στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ορίσει ε, τη διεξαγωγή ενός ε, τραπεζιού εθνικού διαλόγου με όλους τους φορείς ε, για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη χώρα μας, την κοινωνία μας. Περιμένουμε την έκθεση του Οργανισμού Αμερικανικών Χωρών και ο πρέσβης ε, κύριος Σοτσόα, φυσικά θα παρουσιάσει όλα αυτά τα πορίσματα και με κάθε διαφάνεια και τη δική μας τοποθέτηση. Ως ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Ατάλα. Θέλω να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Κοστέλο από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε πρέπει να πω ότι και εσείς και η κυρία Μαρίσα Ματίας εξηγήσατε πολύ καλά τα ε, γεγονότα και την όλη αυτή διαδικασία. Αν μου επιτρέπετε να κάνω εγώ κάποιες πιο γενικές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι είναι σημαντικό πραγματικά να επισημάνουμε ε, τη μεγάλη επιτυχία αυτής της αποστολής εκλογικής παρατήρησης. Έγινε πολύ εντελεχής δουλειά αυτό κάνουμε συνήθω βέβαια στι αποστολέ μα, αλλά πραγματικά ήταν ενδελεχέστατη η όλη παρακολούθηση από την προεκλογική εκστρατεία μέχρι και τι προσφυγέ. Και πρέπει να σα πω ότι αυτό για μα είναι ένα υπόδειγμα ουδετερότητα αμεροληψία σε ό,τι αφορά ε, την εκλογική παρατήρηση, που σημαίνει ότι αυτή η αποστολή εκλογική ε, παρατήρηση και στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή θα έλεγα, όταν υπήρχε και αρκετή εκλογική βία θα έλεγα, η αποστολή και η Μαρίσα είχαν ε, το κύρος και μπορούσαν να συνομιλήσουν με όλους ε, τους εμπλεκόμενου φορεί και για παράδειγμα να πείσουν τα κόμματα της αντιπολίτευση πως έπρεπε να κάνουν τις προσφυγές τους διαμέσου του επίσημου δικαστικού συστήματος και την εκλογική επιτροπή ε, είχαν επικοινωνία για να τις ζητήσουν παράταση της προθεσμίας. Άρα η αποστολή ουσιαστικά κατέβνασε τα πνεύματα γιατί πραγματικά η κατάσταση ήταν πραγματικά πάρα πολύ στα όρια θα έλεγα. Αυτό θέλω να το πω από τη δοσφοροτιμή στη Μαρίσα. Το δεύτερο που θέλω να πω, διδαχθήκαμε αρκετά από αυτή την αποστολή. Η αποστολή εκλογικής παρατήρησης, και μιλώ γενικά τώρα σαν θεσμός, ε, πολλές φορές αντιμετωπίζει ένα επίπεδο επιθέσεων, αν θέλετε, που κατά το παρελθόν δεν είχε να αντιμετωπίσει. Δηλαδή, κατά το παρελθόν ήταν ε, στο πλαίσιο αυτών των εκλογών οι αποστολές εκλογικής παρατήρησης και θεωρούνταν ένας αμερόληπτος ε, παράγων που έπειτα θα επέβαλαν αφόρες. Ε, αυτό βλέπουμε να αλλάζει σε αρκετές περιοχές. Αυτό δηλαδή που λένε δημοσία, αυτές οι αποστολές ε, παρακολουθείτε, ελέγχεται πολύ πιο αυστηρά. Αυτοί που θέλουν να επιτεθούν στην ακερότητα μιας εκλογικής διαδικασίας θα χρησιμοποιήσουν δηλαδή πλέον την αποστολή παρατήρηση και το τι λέει αυτή για να αντιπαραβάλουν αυτά με το αφήγημα που μπορεί να λέγεται στην, άλλη πλευρά Μάθαμε πολλά από τι εκλογέ στην Ονδούρα, γιατί ακριβώ ήταν πάρα πολύ επιτυχής η αποστολή σε αυτό, ότι απέφυγε να τη χρησιμοποιήσουν, να την εκμεταλλευτούν κατά αυτόν τον τρόπο. Ήταν πάρα πολύ εύκολο να είχε συμβεί αυτό και δεν συνέβη και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, σε σχέση με την όλο και μεγαλύτερη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών ε, στι εκλογέ, Αυτό αποτελεί πρόκληση για τι αποστολέ εκλογική παρατήρηση γιατί ο βαθμό τον οποίο, όπω στην περίπτωση τη Ονδούρα, που γίνεται μεταδίδ η μετάδοση συγγνώμη, των αποτελεσμάτων, αλλά και οι υπολογισμοί και τα διάφορα συστήματα, ποιο θα τα λοιπά. Αυτό μπορεί κανείς πάρα πολύ δύσκολα να το παρατηρήσει. Είναι ένα είδος, πώς να το πω, μαύρου κουτιού. Στην περίπτωση της Ονδούρας, όπως ακούσαμε, αυτό το οποίο θα μπορούσε να είναι μια πλήρης καταστροφή το βράδυ των εκλογών, Φαίνεται ότι κατάρρευσε το σύστημα το πληροφορικό και επίσης φάνηκε να αλλάζουν τα αποτελέσματα ε, πριν τη διακοπή δηλαδή της μετάδοσης ε, και μετά ε, και αυτό δημιούργησε φυσικά μεγάλες ε, υποψίες. Αυτό το οποίο κατέβνασε και διασκέδασε τις ε, υποψίες είναι ότι είχαμε εκλογικά τμήματα τα τελικά αποτελέσματα, τα πολιτικά κόμματα είχαν αντίτυπα αυτών των τελικών αποτελεσμάτων, αυτών των πρακτικών. Αυτά ηλεκτρονικά διαβάστηκαν στα κεντρικά και έπειτα δημοσιοποιήθηκε στο διαδίκτυο επίσημη αυτή έκδοχη ας πούμε, των αποτελεσμάτων από τα κεντρικά. Και υπήρχε δυνατότητα σύγκρισης των δελτίων αποτελεσμάτων και αν αυτά δεν φωνούσαν μεταξύ τους ε, μπορούσε να γίνει αυτό, να επαληθευτεί αυτό. Και αυτό επέτρεψε και εξασφάλισε τελικά, πώς να το πω, έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο στην ε, ηρεμία που επικράτησε και ότι διασκεδάστηκαν τελικά υποψίες ότι κάποιοι είχαν εκμεταλλευτεί το σύστημα πληροφοριών. Αντικειμενικές δηλαδή, αποστολές νομίζω ότι ποτέ δεν θα εμπλακούν σε τεχνολογίες πιστοποίησης που σχεδιάζονται για τις εκλογές. Αυτό απαιτεί κάποια συγκεκριμένη εμπειρία και τεχνογνωσία. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αρχίζουμε να ε, μελετάμε αυτά τα μαύρα κουτιά, αν θέλετε. Εμείς ως παρατηρητές. Και για να υπάρχει αυτή η ε, επιτυχία να συνεχιστεί, είναι καλό να υπάρχει ένα ίχνος, ε, πώς να το πω, έντυπο. Να μην έχουμε μόνο ηλεκτρονική διαβίβαση, αλλά να έχουμε να συγκρίνουμε και χαρτιά, τα τελικά αποτελέσματα. Και ένα τρίτο που θέλω να πω σε σχέση με αυτό το εκλογικό σύστημα στην Οδόρα και πώς μπορεί κάπως να μεταρρυθμιστεί για να μην προκύψουν αντίστοιχα φαινόμενα. Είναι καλό να τα δούμε όλα αυτά, αλλά είναι σημαντικό επίσης να πούμε ότι Είδαμε παρόμοιε αδυναμίε με το 2013 στο εκλογικό σύστημα, όπω για παράδειγμα δυσκολίε ε, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των εκλογικών τμήματων και το ρόλο των πολιτικών κομμάτων και επίσης κάποιες ε, υπερβολικές ε, εγγραφές, πλεονάζουσες εγγραφές στα μητρώα εκλογικά. Όταν αποφασίζουμε να πάμε σε μια χώρα για τις εκλογές, αυτό αποτελεί επένδυση δεν μπορεί να πάει σε πολλέ χώρε της Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθεί εκλογέ, άρα για μα είναι όλο και πιο σημαντικό όταν πηγαίνουμε σε μια χώρα και όταν επανερχόμαστε και διατυπώνουμε τι συστάσει μα, αν μα ζητηθεί να παραστούμε και σε επόμενε εκλογέ ως παρατηρητέ, πλέον αρχίζουμε να βλέπουμε σε σχέση με τις συστάσεις που είχαμε διατυπώσει την προηγούμενη φορά, πόσες από αυτές ε, εισακούστηκαν ε, και αυτό είναι και ένα κριτήριο ε, για να αρχίσουμε τις προτεραιότητες μας από κοινού βέβαια με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για μελλοντικές αποστολές εκλογικής παρατήρησης. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Πόνς, αναπληρωτή διευθυντή της αρμόδιας υπηρεσίας της εξωτερικής δράσης για την Κεντρική Αμερική. Έχετε το λόγο. Si bueno muchas Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και αυτά που είπατε εσείς, αλλά και αυτά που είπε η κυρία Ματίες και ο προλαλής σας, εξήγησαν νομίζω πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια ξανά σε όλους όσοι συμμετείχαν στην εκλογική αποστολή παρατήρησης και ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κυρία Ματίας για το εξαιρετικό της έργο κάτω από συνθήκες ιδιαίτερα σκληρές και δύσκολες. Θέλω επίσης να να λάβω τα συλληπιτήριά μας για όλα αυτά τα θύματα μετά τις εκλογές. Εμείς είπαμε ότι και οι δύο πλευρές θα έπρεπε να συμπεριφέρονται υπεύθυνα και όχι να προχωρούν σε δράσεις που αναζωογονούν τις εντάσεις και τις επιθέσεις. Υπήρξε και δήλωση της είπα του εκπροσώπου για ειρηνικές διαδηλώσεις. Εμείς παρακολουθήσαμε τις εκλογές αυτές κάτω από δύσκολες συνθήκε όπως είπαμε, αλλά ήμασταν προετοιμασμένοι να συνεργαστούμε με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές και σίγουρα ε, στηρίζουμε ιδέες όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Πιστεύουμε ότι Μετά από το Σάββατο που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Πρόεδρος, εμείς είπαμε ότι στο μέλλον πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις ώστε το κράτος δικαίου, η διακυβέρνηση, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να λαμβάνουν χώρα όπως πρέπει, όπως επίσης και η σταθερότητα και τα καταπολέμηση της διαφθοράς και της ατιμορρησίας. Χαιρετίζουμε επίσης πρωτοβουλία για διάλογο γιατί Θέλουμε να γίνει ένας διάλογος με συμμετοχή όλων στα σοβαρά και να υπάρξει κάποια διαμεσολάβηση μεταξύ των πλευρών που βρίσκονται σε αντιπαράθεση. Ελπίζουμε επίσης οι εκλογικές μεταρρυθμίσεις να υλοποιηθούν όπως τις συστήνουν οι διάφορες αποστολές και αυτό να βοηθήσει για ένα καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους να ξεκινήσω με τον κύριο Φοντάγνε, όχι, όχι. Δεν θα είμαι δίκαιη. Με τον κύριο Φαρία, μετά ο κύριος Ιτουρκάτς, συγγνώμη είναι πολύ δύσκολο το όνομά σας, και μετά η κυρία Φοντάν. Ευχαριστώ. Ε, muito obrigado, Sr. Presidente. De facto... Ah, já? É o tema. Sim. Pois. <laughs> Ponto para mim. Ehm, <laughs> Ευχαριστώ πολύ. είναι Θέλω να πω, λέει ο κύριο Φαρία, ότι ο επικεφαλή τη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι στην ε, ε, αποστολή με την Βερόνικα Φαντανιέ, τον κύριο Τουγκάη, τον κύριο Χαουρίκη και τον Σέρτζιο Λόπεθ. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, απλώς να πω ότι εμείς πήγαμε εκεί να παρατηρήσουμε την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Όπως είπε και η Μαρίσα, περιοριστήκαμε στην παρατήρηση της εκλογικής διαδικασίας τη συγκεκριμένη μέρα δεν υπήρξαν επεισόδια, δεν υπήρξαν ανομαλίες, υπήρξε διαφάνεια την ημέρα των εκλογών. Τώρα η Μαρίσα εξήγησε τι έγινε πριν και μετά. Και θέλω να προσθέσω μία πληροφορία. Διαπιστώσαμε πέρα από όλη αυτή τη διαδικασία, παρατηρήσαμε πώς εργάστηκαν η Μαρίσα για παράδειγμα, και εδώ θέλω να βγάλω το καπέλο πραγματικά στη Μαρίσα, γιατί η δουλειά που έκανε ήταν εξαιρετική. Σε ένα κλίμα έντασης που το ένιωθε κανείς, το ανέπνε και κατάφερε η Μαρίσα να παίξει έναν πάρα πολύ καλό ρόλο. Ανέλαβε τον ρόλο που της έπρεπε ως πρόεδρος της δικιάς μας ε, ε, αποστολής παρατήρησης των εκλογών, που δεν ήταν εύκολο, το είπα και το ξαναλέω, το διαπιστώσαμε όλοι και διαπιστώσαμε όλοι επίσης ότι υπήρξαν ε, περίπλοκες καταστάσεις που προέκυπταν ε, κάθε τόσο. Παντός έχω συμμετάσχει και σε άλλες ε, τέτοιες αποστολές, αλλά αυτό ήταν κάτι ιδιαίτερο. Γι' αυτό και πάλι λέω μπράβο και συγχαρητήρια στη Μαρίσα και σε όλη την αποστολή, γιατί επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω το έργο τους ήταν εξαιρετικό. Αντίθετα από ό,τι συμβαίνει σε άλλες ε, τέτοιες αποστολές όπου συμμετείχα, εδώ πραγματικά ήταν εντελώς αμερόληπτη η Μαρίσα Ματίας και θέλω να τη συγχαρώ και εκείνη και όλους γιατί πραγματικά μας έβγαλαν ασπροπρόσωπους. Τώρα τα αποτελέσματα πράγματι έφτασαν μετά από τα όσα έγιναν, τα πήραμε εμείς, αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι τα πράγματα έγιναν όπως έπρεπε από τη δικιά μας πλευρά και όπως είπαν και άλλοι και από την Κομισιόν και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, δυστυχώς υπήρξαν μετά ε, συμβάντα με τα οποία χάθηκαν και ζωές. Και αυτό βέβαια αμαυρώνει κάπως την κατάσταση. Αυτά. Η δικιά μας αποστολή, επαναλαμβάνω, ήταν παρατήρησης την ημέρα των εκλογών, όπου εμείς δεν διαπιστώσαμε τίποτα το ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθ' άλλο. Και ξέραμε εξάλλου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπόταν εξαιρετικά από την Μαρίσα Ματίας. Ευχαριστώ. κύριος Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα επίσης, όπως και ο σύντροφος ε, Χωσέ Γνάθιο Φαρίας, να ευχαριστήσω τη Μαρίσα για την ε, δουλειά που έκανε ως επικεφαλής της αποστολής εκλογικής παρατήρησης στην Ονδούρα. Πραγματικά πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τη δουλειά που έγινε εκεί, από όλους τους υπαλλήλους, ε, αλλά πραγματικά και η Μαρίσα διεύθυνε την αποστολή με υποδειγματικό τρόπο. Ε, ήταν πραγματικά καταπληκτικό. Θέλω να ευχαριστήσω ε, και εγώ, όπως είπε ο Χωσέ Ιγνάσιο, ε, για το πόσο ωραία υποδοχή ήταν για την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η φροντίδα που είχαμε. Τώρα θέλω να πω ότι αν θέλουμε να βάλουμε ένα επίθετο, ε, ένα χαρακτηρισμό, μπορούμε να πούμε ότι είναι συναρπαστικές οι εκλογές ε, και μένω σε αυτό. Ε, με την πρόσφατη ιστορική μνήμη γιατί μπορούμε να θυμηθούμε πώς ήταν σε αυτή τη χώρα προηγούμενες εκλογές, εκλογές και τι έχει γίνει έκτοτε. Αυτή τη στιγμή δεν μας εκπλήσει το γεγονός να γίνονται αυτά τα πράγματα που γίνονται στην Ονδούρα. Η πρόεδρος γνωρίζει, θυμάται πώς μας δέχθηκαν ε, στην ε, Ονδούρα. Μιλώ για τους συντρόφους σας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκεί. Αν μιλήσετε ποτέ με εκπροσώπους ε, της Ονδούρας, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι από την αριστερά, από την αντιπολίτευση δηλαδή, εγώ το λέω, για να μην μου πείτε ότι το λέει δεξιά ή το λέει ο κύριος που το έβγαλε από το μυαλό του, γιατί το είπαν και τα μέσα επικοινωνία της Ονδούρα και τα παγκόσμια. Ο κύριο Νασράλα, ο ηγέτη αντιπολίτευση και υποτελικός υποψήφιο, τι λέει, σα τα διαβάζω ε, αυτό λεξί δεν μπορώ να αποκαλύψω με ποιον θα συναντηθώ. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν οριστεί όχι από την Ονδούρα αλλά έχουν έρθει να παρακολουθήσουν την Ονδούρα σε επόμενες εκλογές και μάλλον έχουν πάρει χρήματα και είναι επικίνδυνοι. Θα έχουμε μία συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν, ποιοι ενέχονται, αλλά είναι σοβαρό για να δούμε ποιοι, γιατί αν δούμε ποιοι ε, πήραν τα λεφτά, ποιοι διεθνείς υπάλληλοι, ε, θα καταρρεύσει ένας πύργος από τραπουλόχαρτα που μέχρι στιγμής είναι ε, στέρεος. Αυτά λέει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση λέει δεν έγιναν εκλογές. Και μάλλον αυτά τα λένε πριν γίνουν οι εκλογές. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζαν εμάς τους... Ε, εκλογικού παρατήρηση. Αυτά έχω να πω. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, αλλά ήθελα να το έχετε υπόψη σα και αυτό εσεί. Ω προ τώρα για τι παρατυπίε, ήταν οι διεθνεί παρατηρητέ εκεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, καταγράψαμε και εμεί τα δικά μα. Δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Σε ό,τι αφορά την ημέρα των εκλογών, πρέπει να πω ότι ήταν ήρεμη. Εμεί κινούμασταν ελεύθεροι, ε, χωρί κανένα πρόβλημα. Δεν είδαμε καμία παρατυπία. Τα πολιτικά κόμματα ήταν παρόντα στα περισσότερα εκλογικά τμήματα ε, από τα οποία περάσαμε, ήταν καταγεγραμμένα. Όταν πήγαμε με τα αποτελέσματα πάντα ε, είδαμε ε, ελευθερία, δημοκρατία και απέναντι στους παρατηρητές και στους ψηφοφόρους. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι πριν, κατά και μετά τις εκλογέ, κύριε Πρόεδρε, όλα τα πολιτικά κόμματα, εκπρόσωποι τους με τους οποίους συναντηθήκαμε, όλοι μα λέγανε πόσο σημασία είχε όχι τόσο το αποτέλεσμα στον υπολογιστή, στο σύστημα πληροφορικής, αλλά ε, πόση σημασία θα είχαν αυτά τα δελτία των τελικών αποτελεσμάτων. Άκτας, όπως τα λέμε στα ισπανικά. Δεν ξέρω αν θυμάστε τι έγινε στη Φλόριντα που κέρδισε ο Μπούς τις εκλογές που είχα πιάσει το κάθε ψηφοδέλτιο και το μετράγα γιατί τα πάρα πολύ κοντά οι δύο υποψήφοι. Δηλαδή συμβαίνουν αυτά στις εκλογές. Μπορεί να κρυθεί σε λίγες ψήφους η διαφορά. Έγινε στην ε, Αμερική. Αντίστοιχα πράγματα γίνανε στη δημοκρατία της Ονδούρας. Ε, από τα exit poll, άλλα λέγανε και από τις δημοσκοπήσεις, αλλά τελικά ε, έτσι έγινε. Τα ε, χαρτιά αυτό λένε, ότι ε, κέρδισε αυτός που σήμερα είναι πρόεδρος. Και νομίζω ότι πρέπει να αναγνωριστεί η εκλογική αυτή νίκη. Η δική μας ομάδα, το ΕΛΚΑ, την αναγνωρίζει και χαιρετίζει την νίκη του πρόεδρου Ερνάντες. που ανέλαβε τα καθήκοντά του αυτές τις μέρες, όπως είπε και η κυρία ε, Ματία. Σας ευχαριστώ για το λόγο ε, και για το χρόνο που μου δώσατε. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν έχω να σας πω πολλά, τα είπαν οι συνάδελφοι. Και εγώ θέλω να συγχαρώ, όπως και οι υπόλοιποι, την κυρία Ματίας. Ήταν πολύ καλή πρόεδρος της αποστολής. Από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε και είπαμε ότι η δικιά μας αποστολή ήταν ουδέτερη παρατήρηση εκλογών και είχαμε ό,τι διευκολύνσεις χρειαζόμασταν για να κάνουμε τη δουλειά μας. Όταν πηγαίναμε από το ένα εκλογικό κέντρο στο άλλο, πρέπει να πω ότι η υποδοχή που μας επιφύλασαν τα κόμματα σε κάθε εκλογικό τμήμα ήταν πολύ καλή. Δεν είχαμε πρόβλημα. Ούτε με την καταμέτρηση είχαμε πρόβλημα. Λυπάμαι που τελικά υπήρξαν κάποιες ανομαλίες, αλλά από τη δικιά μου την πλευρά πρέπει να πω ότι για μένα οι εκλογές ήταν σχετικά εκλογές με διαφάνεια και μπορούμε βέβαια να δεχτούμε τη σύσταση ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν ε, στη συνέχεια. Αλλά πάντως υπήρξε ηρεμία την ημέρα των εκλογών. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση από όσα μπορώ να καταλάβω και από όσα άκουσα από τις πληροφορίες, σημαντικές πληροφορίες που μας δώσατε, η αποστολή όντως υπήρξε σημαντική και επιτυχημένη και θέλω να ε, δώσω θερμά συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν σε αυτή. Ήταν υποδειγματική αποστολή, ε, ε, φαίνεται. Ε, αυτό που θέλω να πω και θέλω να καταγραφεί είναι ότι όλοι καταδικάζουμε την βία και κυρίως έχει να κάνει και με απώλειες ανθρώπινων ζώων ότι θα περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα και ότι σαν Επιτροπή τότε θα κάνουμε ξανά μια συζήτηση πάνω στο ίδιο θέμα. Τώρα θα πρέπει να πάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο από ό,τι βλέπω, και αφορά την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την προετοιμασία της επίσκεψης αντιπροσωπείας στο Ελ και την Καράγουα, που την έχουμε ορίσει για τις 12 έως τις 16 Φεβρουαρίου του 2018. Πληροφορίες βρίσκεται στο σχέδιο του προγράμματος φακέλους που σας έχουν διανεμηθεί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στις δύο χώρες, τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν με εκπροσώπους των νομοθετικών οργάνων της κυβέρνησης, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα. Θα ήθελα να σας αναφέρω αναλυτικά με ποιους θα συναντηθούμε, αλλά δεν θα το κάνω ακριβώς για να δώσω περισσότερο χρόνο στους ε, δύο πρέσβεις να μας μιλήσουν για αυτή την αποστολή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η επίσκεψη αντιπροσωπεία παραμένει αβέβαιη λόγω τη χαμηλή συμμετοχή των μελών. Δυστυχώ μέχρι τώρα δύο μονάχα μέλη έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή και θέλω να τονίσω ότι η επίσκεψη με δύο μέλη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Θα δώσω ένα περιθώριο στι πολιτικέ ομάδε να προσπαθήσουν να βρουν περισσότερα μέλη μέχρι την Τετάρτη στο τέλο του εργασιακού ορίου και αν αυτό δεν γίνει εφικτό θα είμαι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένη να αναβάλω την επίσκεψη αντιπροσωπεία για μια άλλη ημερομηνία. Θέλω να επισημάνω επίση ότι οι δικαίωμα συμμετοχή έχουν και τα μέλη τη Eurolat σε αυτή την ε, αποστολή. Τώρα θα μου επιτρέψετε να δώσω τον λόγο στην αυτού εξοχότητα πρέσβη του Ελ τον κύριο Βιλατότο, για να σχολιάσει την επίσκεψη αντιπροσωπεία και να κάνει μια σύντομη εισαγωγή στην ε, τρέχουσα πολιτική κατάσταση του Ελ Σαλβαδόρ. Ευχαριστώ. Muchas eh. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζω και εγώ τους Ευρωβουλευτές ΕΔΕ και τους συναδέρφους πρέσβεις που εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και των ε, αποστολών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα προσπαθήσω να συνοψίσω λίγο κάποια θέματα που εμείς πιστεύουμε ότι έχουν σημασία προκειμένου να γνωρίσετε καλύτερα τι συμβαίνει στο Σαλβαδόρ. Και ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε να έρθω εδώ και να σας μιλήσω για την επίσκεψη αυτή που ελπίζουμε να μην ακυρωθεί. Που θα υπάρξει απαρτία, ελπίζουμε, ώστε να λάβει χώρα. Θα γίνει λοιπόν από τις 12 μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου φέτος, έτσι. Οπότε πρέπει να ξέρετε ότι στο Σαλβαδόρ βρισκόμαστε σε προεκλογική εκστρατεία γιατί 4 Μαρτίου γίνονται οι εκλογές εκεί ώστε να εκλέξουμε δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και βουλευτές στη χώρα μας. Η κοινοβουλευτική συνέλευσή μας έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι υπεύθυνη για την ε, για τον ορισμό μάλλον των δικαστών μας, οι οποίοι θα αναλάβουν τα καθήκατά τους από τον Ιούλιο και μετά. Δέκα κόμματα έχουν εγγραφεί και θα συμμετέχουν με υποψηφίους στις εκλογές αυτές. Και ο Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Γούγκο Μαρτίνες, έχει επεκτείνει πρόσκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να συμμετέχετε κι εσείς με αποστολή παρατηρητών. Έγινε αποδεκτή η πρόσκληση αυτή και ήδη βρίσκονται στο Σαλβαδόρ κάποιοι αξιωματούχοι που προετοιμάζουν την αποστολή αυτή. Ευχαριστούμε πολύ επίσης που δεχτήκατε την πρόσκληση αυτή και που ήδη ε, αναλάβατε κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα υπάρξουν και άλλοι παρατηρητές, όπως για παράδειγμα από τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών, από το Παγκόσμιο Οργανισμό Εκλογών, αλλά και πυρογνώμονες της Λατινικής Αμερικής για θέματα εκλογών. Προβλέπεται επίσης να συμμετέχουν κάπου 2.000 άνθρωποι ως παρατηρητές. Αυτά για τις εκλογές. Από την άλλη, θα μου επιτρέψετε να σας μιλήσω λίγο για το θέμα της άμβλωσης. Και τα σεξουαλικά δικαιώματα των γυναικών στο Ελ Σαλβαδόρ. Όλοι γνωρίζουμε ότι στις 14 Δεκεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το Σαλβαδόρ όσον αφορά τις περιπτώσεις γυναικών που διώκονται επειδή είχαν αποβολή, λέει η ομιλήτρια. Να ξέρετε ότι εμείς το ψήφισμα αυτό το στείλαμε στις αρμόδιες αρχές και όπως καταλαβαίνετε, σε ένα κράτος δικαίου υπάρχουν διάφορα όργανα διαφορετικά και είναι η συνέλευση η οποία τελικά ε, ψηφίζει και αποφασίζει και η νέα της 4ης Μαρτίου θα αναλάβει να παρακολουθήσει και νομοθετικά τα συνταγματικά ζητήματα και το τι θα ισχύει. Οπότε εμείς στείλαμε το ψήφισμα εκεί που έπρεπε, αλλά πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά το κόμμα, ε, το παροντού το Μαρτί, βρίσκεται σε μεταρρύθμιση όσον αφορά τον ε, ποινικό κώδικα, ώστε ακριβώς να αποποινικοποιηθεί η άμβλωση. Εφόσον κινδυνεύει η ζωή της ε, μητέρας πρώτον, δεύτερον εφόσον η εγκυμοσύνη οφείλεται σε βιασμό, τρίτον όταν υπάρχει δυσμορφία στο έμβριο και τέταρτον σε περιπτώσεις που βρίσκεται υπό ναρκωτικά κλπ. Να ξέρετε ότι εγώ μαζί με όλους τους υπόλοιπους κάνουμε προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων της γυναίκας εφόσον βρίσκεται σε κατάσταση όπως ε, σε εγκυμοσύνη μετά από βιασμό ή οτιδήποτε άλλο που να δικαιολογεί τελικά την άμβλωση. Υπάρχει πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται στο Σαλβαδόρο σήμερα εδώ και πέντε χρόνια που προστατεύει τη γυναίκα και ακριβώς η Προεδρία της χώρας θέλησε να έχει αυτό το πρόγραμμα για να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες μέσω ειδικευμένων υπηρεσιών για να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους, για να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες που ε, τους προσφέρουμε κλπ. Το πρόγραμμα αυτό που ονομάζεται Ciudad Mujer περιλαμβάνει την υγεία, την απαραγωγική και τη σεξουαλική, δεύτερον την βία σε βάρος των γεγονών, την αυτονομία την οικονομική και ε, την ε, προσοχή στα παιδιά. Τώρα με την ε, επίσκεψη που θα κάνετε, για την προσωπία σας δηλαδή, αν αυτή όντως λάβει χώρα, να ξέρετε ότι προβλέπουμε και επίσκεψη σε ένα από τα κέντρα αυτά που υπάρχουν στο Σαλβαδόρ με το πρόγραμμα αυτό Ciudad Mujer. Έχει μεγάλη επιτυχία και που στηρίζεται το πρόγραμμα αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βασική ιδέα του προγράμματος αυτού είναι οι γυναίκες να έχουν περισσότερη εξουσία και να μπορούν να αναλάβουν τη ζωή τους και να πάρουν αποφάσεις για τη ζωή τους, να έχουν οικονομική αυτονομία και βέβαια να μην ε, υποφέρουν από αδικογενειακή βία. Κάτι άλλο σημαντικό για τη χώρα μας και το ξέρετε όταν ήρθε ο Γκομαρτίνες ε, εδώ, Ξέρετε για το άλλο μας το πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Ασφαλές El Salvador. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια. Η κυβέρνηση στη χώρα προσπαθεί όσο γίνεται καλύτερα να αντιμετωπίσει το θέμα της ασφάλειας στη χώρα. Το ξέρετε αυτό το πρόγραμμα και επιτρέψτε μου λίγο να σας πω τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα με το πρόγραμμα αυτό. Για παράδειγμα, το 2017 μειώθηκαν σε ένα μεγάλο βαθμό, κατά 27% δολοφανίες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Επίσης, μειώθηκαν πάρα πολύ στους 10 δήμους οι δολοφονίες εκεί όπου ακριβώς εφαρμόζεται το πρόγραμμα, σε 50 δήμους δηλαδή. Τώρα έχουμε περάσει στο τρίτο στάδιο που περιλαμβάνει και τους 24 δήμους που δεν συμμετείχαν μέχρι τώρα. Υπάρχει λοιπόν σαφώς βελτίωση όσον αφορά την πρόληψη της βίας σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο μέσω θεσμικών δομών από το αρμόδιο Υπουργείο και έχουμε προχωρήσει σε προγράμματα εκπαιδευτικά προκειμένου να μπορέσουμε να επανεντάξουμε σε εκπαιδευτικά συστήματα ανθρώπους οι οποίοι είχαν μείνει εκτός, ομάδες που είχαν ε, βρεθεί στη βία και έτσι με το πρόγραμμα αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Τώρα γίνεται η αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος ε, αυτού, πια επίσημα, για να μπορέσουμε να δούμε αν χρειάζεται κάποια βελτίωση. Είναι βέβαιο όμως ότι τα ωφέλη είναι πολλά για το Σαλβαδόρ μέχρι τώρα. Κάτι άλλο το οποίο μας ε, ενδιαφέρει είναι η Συμφωνία Σύνδεσης που ενδιαφέρει και την Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια. Προς το παρόν, όπως όλοι γνωρίζουμε, ισχύει μόνο το εμπορικό σκέλος και όχι ο πολιτικός πυλώνας και συνεργασίας. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε έκκληση για άλλη μια φορά προκειμένου να υλοποιηθεί και αυτό το σκέλος και να υπάρξει πλήρη κύρωση της συμφωνίας αυτή. αυτής. Προς το παρόν, μόνο τέσσερις χώρες παραμένουν χωρίς ε, να έχουν προβεί στην κύρωση και τα ωφέλη από την εφαρμογή, ε, την αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας αυτής είναι τεράστια. Οι προσδοκίες του Ελσαλβαδόρ είναι πολύ μεγάλες και φέτος θα θέσουμε σε εφαρμογή διάφορες δράσεις προκειμένου να δώσουμε νέο δυναμισμό στην εφαρμογή της συμφωνίας αυτής σύνδεσης, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών. Τέλος, όπως όλοι γνωρίζουν, έχουμε την Προεδρία προσωρινά της ΕΛΑΚ. Και με ιδιαίτερη χαρά μπορώ να σας πω ότι πρόσφατα κάναμε ανακοίνωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζοντας την επιθυμία μας να βρεθεί μια ημερομηνία όπου θα μπορέσουμε να έχουμε η Υπουργική Συνεδρίαση Υπουργών Εξωτερικών σε ΛΑΚ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι που περιμένουμε και συνεργαζόμαστε ώστε να βρεθεί η ημερομηνία αυτή, ώστε φέτος να υλοποιηθεί η συνάντηση αυτή και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε και ελπίζουμε επίσης να έχουμε και τη δικιά σας στήριξη όπως την πήραμε από άλλες περιφέρειες. Αυτά, τίποτα άλλο. Όλα αυτά έχουν αποφασιστεί από το Υπουργείο Εξωτερικών όσον αφορά τη ΣΕΛΑΚ, έκτακτη συνεδρίαση που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα και το Ελ εξακολουθεί προσωρινά να έχει την Προεδρία της ΕΛΑΚ. Γι' αυτό να ξέρετε ότι είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με επιτυχία όπως το κάναμε και μέχρι τώρα. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ κυρία Πρέσβη. Ήσασταν χήμαρο όσα μα είπατε, πολύ σημαντικέ πληροφορίε που μα δώσατε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σαντίνο να μα κάνει και εκείνο κάποια σχόλια για το επικείμενο ταξίδι, αλλά και να μα πει για την πολιτική κατάσταση στην Καράβο σήμερα. <clears throat> Σα ευχαριστώ πολύ, αξιότιμη Σοφία πρόεδρε τη ΔΕΚΑΜ, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, συνάδελφοι, αξιότιμοι πρέσβει, εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή και τη ΕΙΕΔ, φίλε και φίλοι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Δανίλη Ορτέγα και αντιπρόεδρος σας στέλνουν ευγενή χαιρετισμό. Πρόκειται για πολύ μεγάλη χαρά για μένα προσωπικά να βρίσκομαι εδώ ξανά. Ήμουν εδώ στις 4 Δεκεμβρίου, οπότε και σας παρουσίασα μία έκθεση σε σχέση με τις δημοτικές εκλογές στην Καράγουα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι ο πρόεδρος Ορτέγα συνεχίζει να χαίρει ευρύτατης λαϊκής υποστήριξης 80% περίπου των κατοίκων της Νικαράγουας εξέφρασαν την κανοποίησή τους προς την κυβέρνηση. Και βέβαια ενισχύεται με τον τρόπο αυτό η αισιοδοξία και υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και των ξένων παραγόντων και ξένων επενδυτών στη χώρα μας. Παίξα ένα ρητό αίτημα και πρόσκληση από την ΤΕΚΑΜ για να ξαναέρθουμε σήμερα εδώ και για να σας παρουσιάσουμε την κατάσταση, κυρίως την οικονομική κατάσταση της χώρας και βέβαια ελπίζουμε ότι στην επίσκεψή σας που μακάρι να λάβει χώρα μεταξύ 14 και 16 θα πάρετε πολύ περισσότερες πληροφορίες. Πρέπει να σας πω ότι το οικονομικό μοντέλο που υλοποιούμε στην Ικαράουα στόχο έχει να ανταποκριθεί σε δύο απαιτήσει. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε να δημιουργήσουμε ε, αγαθά και να τα αναδιανύμουμε με δίκαιο τρόπο και θέλουμε να έχουμε βέβαια στο δυνατόν ε, μεγαλύτερο δημόσιο όφελος για τους πολίτες. Έχουμε το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο το οποίο έχει ήδη κατατεθεί και το γνωρίζει η κοινωνία της ε, Νικαράγουας. Ο στόχος μας είναι να προωθήσουμε τις δεξιότητες, ε, την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και να αναπτύξουμε τα απαραίτητα συστατικά για την ανάπτυξη στην Νικαράγουα με βάση τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της χώρα μας για το 2017 η ανάπτυξη ήταν της τάξης του 5,2%. Κάτι το οποίο θεωρείται πολύ θετικό, όπως επάλ βλέπουμε δηλαδή αύξηση Επίσης και των ε, εξαγωγών μειώνεται σιγά σιγά ε, το έλλειμμα το εσωτερικό. Καταφέραμε λοιπόν να μειώσουμε ε, το έλλειμμα αυτό σε 8% και έτσι μπορούμε να έχουμε περισσότερα έσοδα, έχουμε 10% αύξηση των κοινωνικών εμβασμάτων και πολύ καλή ε, κίνηση τουριστική, αύξηση 30% ε, για τον τουριστικό κλάδο. Σε ό,τι αφορά την προσφορά της εργασίας στη χώρα μας, είχαμε και εδώ αύξηση 5,7% περισσότερα άτομα είναι καταχωρημένα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, που σημαίνει ότι προοδεύουμε και στον τομέα αυτό καταπολεμούμε την επισφαλή εργασία. Για το 2018 στόχος μας είναι να παραμείνουμε σε αυξητικές τάσεις και έτσι προβλέπεται 1,5% ο δε πληθωρισμός μεταξύ 5 και 6,6%. σχετικά ελεγχόμενα, δηλαδή τα επίπεδα. Με τον τρόπο αυτό πιστεύω θα εξασφαλίσουμε και τη σταθερότητα των τιμών για το 2018. Σε ό,τι αφορά εξωτερικέ ροέ. Ελπίζουμε να υπάρξει αύξηση 1,4 δις δολάρια σε ό,τι αφορά τα project, σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές και έχουμε και το διάλογο, συμμαχία και συνένεση μεταξύ ιδιωτικού δημόσιου τομέα και ε, συνδικάτων. Αυτή η διαδικασία στηρίζει την σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη, Είναι πολύ σημαντική διαδικασία. Πρέπει να σας πω ότι διεθνώς αναγνωρίζεται αυτός ο εθνικός διάλογος και η σημασία του, διότι πραγματικά εδραιώνει την εμπιστοσύνη και βελτιώνει το επενδυτικό κλίμα. Τώρα, πολιτική κατάσταση. Υπήρξαν διάφορες εκλογές με βάση το εκλογικό χρονοδιάγραμμα. Εργαζόμαστε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών με στόχο την ενίσχυση και βελτίωση του δημοκρατικού συστήματος της χώρας. Τέλος, θα ήθελα να κάνω κάποια γρήγορα σχόλια σε σχέση με το θέμα της ασφάλειας. Λόγω της γεωγραφικής μας θέσης έχουμε ε, δραστηριότητα ε, λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Είναι ένας ε, τόπος διέλευσης δυστυχώς η χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια Καταφέραμε όμως ε, να ε, ανεγείρουμε, αν μπορώ να το πω, ένα τείχος συγκράτησης ε, αυτών των κινήσεων και της διακίνησης ναρκωτικών. Και έχουμε ξαναπεί ε, τις πρόοδος που έχουν επιτευχθεί στην Επιτροπή σας, στην αντιπροσωπεία σας και ελπίζουμε και εσείς να Θελήστε να διανύμετε, έχουμε κάποια στοιχεία, αν θέλετε μπορείτε να τα διανύμετε σε όλους τους συναδέλφους σας. Η Νικαράγουα υιοθετεί ένα κοινοτικό και προληπτικό σύστημα προστασίας των πολιτών για την προστασία ατόμων, ε, οικογενειών ε, και κοινωνιών εν γέννη ώστε και οι πολίτες με τη συμμετοχή τους ε, να μπορούν να βελτιώνουν ε, αυτό το μοντέλο το κοινωνικό και να ζουν σε συνθήκες ασφάλειας. Ελπίζω να μπορέσετε να επιβεβαιώσετε αυτό το μοντέλο ε, όταν έρθετε στη χώρα μας. Θα σας περιμένουμε και θα δείτε τη φιλοξενία που μπορούμε να σας παράσχουμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πόνς, θα θέλετε να πάρετε το λόγο να μας πείτε να μας κάνετε κάποια σχόλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στην αντιπροσωπεία σα για την πρωτοβουλία να επισκεφτείτε αυτέ τι δύο χώρες. Δύο χώρε που και οι δύο είναι δυνατοί εταίροι μα. Για να ξεκινήσω με το Ελσαλβαδόρ, οι σχέσει μα είναι εξαιρετικέ ο Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Μαρτίνε, ήρθε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τον Απρίλιο που μα πέρασε και μάλιστα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήρθε και σε εσά, στην αντιπροσωπεία σα, σε μια εκείνη συνεδρίαση που έγινε και όπου τέθηκαν πολλά και διάφορα θέματα. Χαιρόμαστε πολύ με την απόφαση του Ελσαλβαδόρ να συμμετέχει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και με ικανοποίηση επίσης παρατηρούμε την παρουσία του Ελσαβανδόρου στη ΣΕΛΑΚ κάτω από συνθήκες δύσκολες. Μετά από τις παρατηρήσεις της κυρίας Πρέσβος, να ξέρετε ότι ναι, δουλεύουμε για να βρούμε μία ημερομηνία ώστε να λάβει χώρα υπουργική τον Ιούλιο κατά πάσα πιθανότητα. Δουλεύουμε για αυτό το ζήτημα λοιπόν. Επίσης γνωρίσουμε και τις προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπο το Ελσαλβαδόρ. Ανασφάλεια για τους πολίτες. Να ξέρετε ότι φυσικά και στηρίζουμε το πρόγραμμα του Ελσαλβαδόρ για την ασφάλεια των πολιτών και ξέρουμε ότι υπάρχει πρόοδος, αλλά πιστεύουμε ότι σε αυτό το δρόμο πρέπει να προχωρήσει το Ελσαλβαδόρ περισσότερο, προστατεύοντας ε, τα δικαιώματα ακόμα και των ανθρώπων που κάνουν παραβάσεις. Ελπίζουμε να γίνει αυτό, να υπάρξει περισσότερη συνειδητοποίηση. Ε, πρόκληση υπάρχει και όσον αφορά τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Ναι, το γνωρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρουμε ότι γίνονται κάποια θετικά βήματα. Πάντω η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξέρετε ότι θα είναι στο πλευρό σα για να στηρίξει τι μεταρρυθμίσει σα και ότι ε, πρόοδο επιτευχθεί σε αυτό το τομέα όπω πρέπει. Έρχομαι τώρα στην Νικαράγουα. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα στάδιο ιδιαίτερα θετικό όσον αφορά τις σχέσεις μας. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη προσέγγιση. Η υπογραφή συμμετοχή της Νικαράγουα, για παράδειγμα, το, στη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Είναι κάτι που διαπιστώνουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Όπως επίσης και το τι γίνεται όσον αφορά τις δημοτικές εκλογές που έγιναν τον Νοέμβριο και διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν. Υπάρχει διάλογος με την κυβέρνηση της Νικαράγουα, με τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών και πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν ακόμα περισσότερες βελτιώσεις που να είστε σίγουροι ότι θα στηρίξουμε. Συνοψίζοντας λοιπόν για άλλη μια φορά, χαιρόμαστε πολύ που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επισκεφτεί αυτέ τι δύο χώρε. Αξίζει το κόπο και εμεί έχουμε δουλέψει πολύ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να στηρίξουμε αυτέ τι δύο χώρε. Ευχαριστώ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φαρία που θέλει να κάνει κάποια σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να μιλήσω για τις παρανομιακές σχέσεις μεταξύ της Νίκαράγουας και του δικτατορικού καθεστώτος ε, της Βενεζουέλας δεν θα μπορέσω να συμμετάσχω στην αντιπροσωπή αυτή. Μακάρι να πήγαινα στο Ελσαλβαδόρ, κυρία Πρέζη. Δυστυχώ δεν μπορώ εγώ να έρθω στη χώρα σα. Ελπίζω κάποια στιγμή στην προσεχή επίσκεψη για τι εκλογέ στο Ελσαλβαδόρ να μπορέσω να είμαι εκεί. Είναι μια χώρα που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα υπέροχο λαό. Η υποδοχή του είναι καταπληκτική και θα ήθελα να συγχαρείτε την κυβέρνησή σας και να την ευχαριστήσετε που προσκάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο για ε, να συμμετάσχει στην αποστολή εκλογικής παρατήρησης της χώρας σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Φαρία. Θέλει κάποιος άλλος να κάνει κάποιο σχόλιο. Όχι. Θέλετε να... Κύριε Πρέσβη, κυρία Πρέσβη, θέλετε να δευτερολογήσετε. Bueno, brevemente... Ε, ναι, σύντομα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φαρέας για τα πολύ καλά του λόγια και φυσικά ε, με μεγάλη χαρά θα περιμένουμε την επίσκεψή την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, οπότε και θα διεξαχθούν οι εκλογές. Συνάδελφοί σας έχουν ήδη έρθει στη χώρα μου. Α, ήσασταν κι εσείς τότε, α. Μάλιστα, ε, στην Τελάτα. Ε, και επομένως την ξέρετε τη χώρα. Πράγματι η υποδοχή που επιφυλάσσουμε στους επισκέπτες είναι θερμή και όπως είπε και ο πρόσωπος πράγματι υπάρχει θέμα ασφαλείας, αλλά φυσικά και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε η κατάσταση αυτή να μην δημιουργήσει κανένα πρόβλημα και να μην ε, ε, περιορίσει τις κινήσεις ε, των μελών της αντιπροσωπείας. Το θέμα της ασφάλειας είναι πράγματι πολύπλοκο. Παρ' όλα αυτά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά και εσάς προσωπικά κυρία Σακοράφα αλλά και την αντιπροσωπεία σας για τη δυνατότητα που μου δώσετε να είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρέσβη, θέλετε να πείτε. Όχι. Κύριοι συνάδελφοι, έχουμε τελειώσει και με αυτό το σημείο της σημερίσης διάταξης. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ελπίζω να γίνει αυτό το ταξίδι. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται στα σκαριά και γίνονται. Θέλω να πω και στους δύο και στον κύριο Σαντίνο, με τον οποίο έχουμε πάρα πολλές φορές συναντηθεί στην Επιτροπή, αλλά και στην κυρία Βιλατότο, ότι και η Επιτροπή μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριζε και τις δύο χώρες και τις μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να γίνουν. Θέλω να ελπίζω ότι πριν τελειώσει η θητεία μας το θέμα της ολοκλήρωσης της ε, σύνδεσης, ε, της συμφωνίας σύνδεσης θα έχει τελειώσει και να πάμε στο τελευταίο σημείο που πρέπει να ανακοινώσω και να κλείσουμε τη συνεδρίασή μας εκτός και αν υπάρχει κάποιος που θέλει να συμπληρώσει κάτι και συνάδελφοι αν έχετε κάτι να... σαν σχόλιο. Όχι ότι η επόμενη συνάντηση αντιπροσωπείας μας θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου του 2018 στις Βρυξέλλες. Να επαναλάβω τις θέσεις Προεδρίας να οργανώσει για την επόμενη δεκά μια εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων που θα εστιάζει στη δυναμική και στις αναπτυξιακές και επενδυτικές προοπτικές εν ώψη της εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω να συμμετέχετε όλοι σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω θα είναι μια πολύ καλή συζήτηση και θα έχει πάρα εξαιρετικά συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν παρόντες. Ευχαριστώ όλους σας και σας χαιρετώ μέχρι την επόμενη συνεδρία. Να ευχαριστήσω και τους μεταφραστές μας για την βοήθεια που μας παρέχουν κάθε φορά.